και κύριοι, ε, άρχεται η συνεδρίαση και το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η δήλωση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον απολογισμό της Δανικής Προεδρίας και θέλω να χαιρετήσω την απερχόμενη